Προχωρούμε στην ψηφοφορία κυρίε και κύριοι. Το λόγο έχει ζητήσει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ επί διαδικαστικού. Έχετε ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού, κυρία Κοράτσα Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, έχει περάσει πάνω από μήνας από τότε που εδώ στο Κοινοβούλιο αποκαλύφθηκε η εκλογική απάτη, ή ε, μάλλον η μαλλον η απατηση ως προς την ψηφοφορία της κυρίας Λεπέν. Ε, διεξάγετε εσείς μια έρευνα. Θα θέλαμε να ξέρουμε, να γίνει ένας απολογισμός πεπραγμένων, κυρίως για τον κύριο Δεκράφε από την Ευρώπη των Εθνών και για τον κύριο Νίκο Λεμπέη που είναι Γενικός Γραμματέας ε, του Λαϊκού Μετόπου. Θα ήθελα, Πρόεδρε, επίση να σας ρωτήσω εάν προτίθεστε να προσκαλέσετε σε ακρόαση ε, την κυρία Λεπένε, διότι είναι συμπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Ευρώπης των Εθνών και Ελευθεριών. Ευχαριστώ. Ε, Ο πρόεδρος Σούλτς. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Για την παράτυπη και εσφαλμένη αυτή η ψηφοφορία έχω διεξαγάγει έρευνα. Πρώτα για την περίπτωση Δεγκράφ. Άκουσα τον κύριο Δεγκράφ ο οποίος αναγνώρισε ότι δεν ήταν ορθός ο τρόπος που ψήφισε. Τώρα καλούμε να αποφασίσω σχετικά με κάποια κύρωση. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη πια. Θα επιβάλλω κύρωση. Ο κύριος Δεγκράφ μου ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει το ότι ε, ήταν εσφαλμένος ο τρόπος με τον οποίο ψήφισε και ότι θα δεχθεί την κύρωση. Μίλησα και με τον κύριο Αμπέ, ο οποίος σχετικά με την μομφή που απίφθηναν πολλοί συνάδελφοι ότι ψήφισε για λογαριασμό της κυρίας Λεπέν, αυτήν την αρνείται. Δηλώνει ότι δεν το έπραξε αυτό. Μετά από την δήλωσή του αυτή, και επειδή υπήρχαν συνάδελφοι που μου έγραψαν ότι είδαν να το πράττει, παρακάλεσα λοιπόν να προσέλθουν για να συζητήσουμε. Διεξήχθη συζήτηση αυτή, μεταξύ αυτών ε, καταλέγεστε και εσείς ίδια, σας άκουσα και εσάς. Όλοι λοιπόν οι συνάδελφοι αυτοί με διαβεβαίωσαν με πρακτικό υπογεγραμμένο ότι εμένουν, επιμένουν δηλαδή ότι είδαν ότι ο, ο συνάδελφος αυτός ψήφισε με τον τρόπο που περιγράφουν. Θα ξανασυζητήσω με αυτό και θα λάβω τελική απόφαση διότι έχουμε ενώπιό μας μια κατάσταση όπου ορισμένοι 4 5 συνάδελφοι λέγουν ότι τον είδαμε να ψηφίζει, ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος λέει όχι, δεν ψήφισα. Η έρευνα σχετικά με την ε, βουλευτή Λεπέν μου είπαν ότι η κυρία Λεπέν ήταν παρούσα στην αίθουσα. Πρέπει να ακούσω λοιπόν και την κυρία Λεπέν για να μου δηλώσει αν γνώριζε ότι ψήφισε για λογαριασμό τη ο κ. Σαμπέ ή όχι. Το ότι είναι τώρα γραμματεα του ε, Εθνικού Μετώπου δεν παίζει κανένα ρόλο. Όταν θα ολοκληρωθούν όμω οι έρευνε θα, σας, θα προβώ σε σχετικές ανακοινώσεις. Ορίστε εσείς. Είχα, ο κύριος Κράμερ, επειδή ήταν πάρα πολύ μικρή διαφορά του αποτελέσματος, είχα ρωτήσει αν η μία ψήφος έπαιζε ρόλο. Σε διάφορες ψηφοφορίες μάλιστα, όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή πλειοψηφία ή μειοψηφία και η οποία ενδεχομένω προέκυψε μόνο μέσω αυτής της απάτης. απάτης του πρόεδρου Σούλτς. Εξέτασα την υπόδειξή σας, σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει πολύ μικρή πλειοψηφία ή μειοψηφία. Εκεί δηλαδή όπου ψήφισαν οι κύριοι Δεγκράφ ή ε, Αμπέ για λογαριασμό της κυρίας Λεπέν. Σε καμία από τις ψηφοφορίες αυτές δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα εάν είχε ψηφίσει διαφορετικά ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Στην περίπτωση αυτού βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική κατάσταση. Κύριε Γκολνής, ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι παλαιός εδώ. Ο προστάτης μου αυξάνεται όσο μειώνεται η ενέργεια. Ε, εκείνη την ημέρα η ψηφοφορία κράτησε δυόμιση ώρες. Μπορείτε να μου πείτε ε, σε ποιο σημείο ο κανονισμός επιτρέπει η πολιτική παρουσία να διασφαλίζεται ε, παρά τις απαιτήσεις ε, τις σωματικές ή μήπως θα πρέπει να ικανοποιήσω τις σωματικές μου ανάγκες ε, ε, καθήμενος στην έδρα μου. Να θυμίσω επίσης ότι στο παρελθόν στην ε, Γαλλική Εθνική Εθνοσυνέλευση είχα παρατηρήσει την κυρία Τροτμάν, σοσιαλίστρια, που είχε ψηφίσει για πάνω από 160 απόντες βουλευτές με έναν μόνο συνάδελφό της στρέφοντας την κλίδα με παράνομο τρόπο αντίθετα με αυτά τα οποία προβλέπει ο κανονισμός της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης όπως επίσης και του Οργανικού Νόμου και του Γαλλικού Συντάγματος φυσικά. Yeah. Αξιότιμε ε, κύριε συνάδελφε, αξιότιμε κύριε Γκόρνης. Η διαδικασία γύρανσης για όλες και όλους μας είναι μια δύσκολη περίπτωση και μάλιστα φύγει όλα τα όργανα από το κεφάλι μέχρι το πόδι. Έτσι λοιπόν αξίζει πράγματι με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε. Θα συζητήσω ξανά με τις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες για το θέμα σας. Παρακαλώ εσείς κύριε Τόιρερ. Παρετήστε κύριε Τόιρερ. Καλώς. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την ίδρυση ειδική Επιτροπής για φορολογικές συμφωνίες. Σας έχει υποβληθεί η απόφαση του Προεδρείου και πρόκειται για ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το αίτημα, λαμβάνεται η απόφαση δηλαδή, άρα εγκρίνεται η ίδρυση της Επιτροπής και οι σχετικοί διορισμοί. Ερχόμαστε τώρα στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Λίχτενστάιν. Α, με συγχωρείτε, ορίστε. Προβλέπονται δύο ψηφοφορίες στην λίστα. Μία για την ίδρυση και μία για τον διορισμό. Είναι λάθος αυτό. Κοιτάξτε. Διακόπτει ο πρόεδρος. Μια στιγμή, μια στιγμή. Η ψηφοφορία ήταν σωστή. Ο διορισμός ακολουθεί την ψηφοφορία. Άρα λοιπόν σωστός, σωστά πράξαμε. Έκθεση Λούνες. Πρόκειται για ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Λίχτενστάιν για φορολογικά θέματα. Πολύ σωστό άλλωστε μετά από την προηγούμενη ψηφοφορία, αυτή εδώ ακολουθεί. Αρχίζει λοιπόν η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρα. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έρχομαι στην έκθεση των κυριών Μετσόλα Κέλλερ, τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο, παράγραφος 3, υπέρ, κατά, αποχές. Εδώ χρειάζεται επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση επομένω. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 4 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Επαλήθευση. Για πιο σίγουρα. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Σε 5 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Σε τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 12 σε τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 18 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 19 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 21 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, επιθυμείτε επαλήθευση. Επαλήθευση λοιπόν ηλεκτρονική για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε, τέλος. Α, απερίφθη. Οκ. Okay. Παράγραφος 23. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτο, ε, δεύτερο τμήμα, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ θα χρειαστεί επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. εγκρίνεται. 28. Δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 30. Υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση. Αρχίζει η επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η παράγωση 30 λοιπόν. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι υπερψηφίζεται, αλλά θέλετε επαλήθευση. Καλώς λοιπόν. Αρχίζει η επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας 4 δύο πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές λίγο δύσκολο να μορφώσει κανείς άποψη. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. L, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση, καλώς. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Όμικρον, υπέρ, Πρώτο τμήμα δηλαδή κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτό. Θέλετε επαλήθευση. Καλά λοιπόν. Δεύτερο τμήμα ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα αιτιολογική σκέψη Q υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι διαμορφώνει η ίδια πλειοψηφία αν θέλετε όμως επαληθεύω αρχίζει η επαλήθευση τέλος εγκρίνεται ερχόμαστε το τροποποιημένο ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Η έκθεση εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Ντελή για την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Παράγραφος 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Ονομαστική. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20 ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25. Το ίδιο με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 28. Δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, πάλι ονομαστικά, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Σε τρία τμήματα. Ονομαστικά πάντα. Τρία τμήματα αρχίζει πέρας εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα πάλι ονομαστικά αρχίζει ψηφίσατε πέρας εγκρίνεται τρίτο τμήμα ονομαστικά αρχίζει πέρας Εγκρίνεται και αυτό. Το τμήμα, παράγραφος 36, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 39, αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική, αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική, Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 44. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει, τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 45, τροπολογία 1 ονομαστικά. Α, με συγχωρείτε. Κάποιος ζητεί το λόγο. Ορίστε κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τροπολογία που ετοιμάζεστε να ψηφίσετε είναι πάρα πολύ σημαντική. Παρά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της Volkswagen, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν επιδοτήσεις προσωρινά καύσιμα και αναφέρομαι στο ντίζελ που έχει φορολογικά πλέον πλεονεκτήματα και απαλλαγές σε σχέση με τη βενζίνη. Αν θέλουμε να μειώσουμε λοιπόν την χρήση των αυτοκινήτων με τέτοιου είδους ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να δράσουμε. Γι' αυτό προτείνουμε λοιπόν μέσω αυτής της τροπολογίας να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να τελειώνουμε με τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν ήταν διαδικαστικό αυτό. Ήταν ομιλία πολιτικού χαρακτήρα. Εξαρτάται δηλαδή από τα κέφια μα ε, τι δεχόμαστε και τι δεν δεχόμαστε. Διαδικαστικό πάντω δεν ήταν. Πολιτική δήλωση αυτό, το σχόλιο τη κυρία Νταλή. Ο πρόεδρο Σούλτ είναι εισηγήτρια η κυρία Ντελή, ε, κύριε συνάδελφε, και έχει το δικαίωμα να ζητήσει το λόγο. Βέβαια, αν... Διακόπτει ο Βέβαια, κατά αυστηρή ερμηνεία του κανονισμού, οφείλω να της δώσω το λόγο, όχι βεβαίως για πολιτική δήλωση. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλευτήκατε με επιδέξιο τρόπο, κυρία Ντελή, τον κανονισμό. Τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 46, ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία, ψηφίσατε, πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφο 47. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει και τελειώνει. Εγκρίνεται. Άρθρο 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ χρειάζεται επαλήθευση. Ηλεκτρονικά δηλαδή. Αρχίζει, τελειώνει. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η υπαριθμόν 50 ονομαστικά. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 58 ονομαστικά. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 60 ονομαστική. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 62. Πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη κάπα, ονομαστικά. Υπέρ, κατά, α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, παρασύρθηκα. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Υπέρ πάντως 512 κατά Τρεις και έξι αποχές. Αιτιολογική σκέψη μη. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται δε. Και τώρα η αιτιολογική σκέψη Β. Επίσης ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη W. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πάλι ονομαστικά. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 6 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα πάλι ονομαστικά. Ψηφίσατε. Πέρας. εγκρίνεται. Τέλος, το ψήφισμα στο σύνολό του, ονομαστική ψηφοφορία, η οποία αρχίζει, ψηφίσατε, τέλος, εγκρίνεται.